Ε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Καταρχήν καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ θερμά να καθίσετε για να περάσουμε στη ψηφοφορία. Θα ήθελα με ιδιαίτερη χαρά να σας ενημερώσω, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ, λίγη υπομονή και καθίστε για να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Και πάλι λοιπόν να πω ότι με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι η αντιπροσωπεία μας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση για την Ένωση για τη Μεσόγειο θα συναντήσει σήμερα τον κύριο Αντέλ Αλασούμι, αντιπρόεδρο της Αραβικής Βουλής και τον κύριο Αχμέτ Μεσεργή, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Ασφάλειας. Θα ήθελα να εκφράσω ένα θερμό καλωσόρισμα προς τους κυρίους Αλασούμι και Μεσεργή και επευκαιρία να τονίσω τη σημασία που δίνουμε στην αγαστή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Αραβική Βουλή. Καλώς ήρθατε κύριοι Αλασούμη και Μεσέργη. Για διαδικαστικό ε, έχει ζητηθεί ο λόγος, αλλά τονίζω ότι θα δεχθώ τα διαδικαστικά σας σχόλια μόνο εφόσον παραθέτεται και το αντίστοιχο άρθρο του εσωτερικού κανονισμού. Είδε όχι. Ο κύριος Βάγκνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα συμφωνείτε ότι είναι σημαντικό αυτό το θέμα και θέλω να πω δύο λόγια. Ε, νομίζω ότι ένα διακόπτει ο πρόεδρος. Δεν είναι διαδικαστικό αυτό. Δεν αναφέρατε κανένα άρθρο του εσωτερικού κανονισμού. Είπα ότι θα δεχτώ τα σχόλια για διαδικαστικά ζητήματα μόνο εφόσον συνοδεύονται από ε, άρθρα του εσωτερικού κανονισμού. Έχουμε ένα ε, μεγάλο αριθμό σημαντικών νομοθετικών θεμάτων. Πρέπει να τα διεκπαιρεώσουμε στις ψηφοφορίε. Η κυρία Γκόμες, τι διαδικαστικό έχετε. Ο κύριο Μερέρα Κοντίνα αποφυλακίστηκε στην Αιθιοπία. Εμεί ζητήσαμε την αποφυλάκησή του και επιτέλου απελευθερώθηκε. Καλώ το σημειώνουμε, αλλά περάσουμε παρακαλώ στις ψηφοφορίε, γιατί δεν ήταν διαδικαστικό ούτε το ένα ούτε το άλλο σημείο. Κυρίε και κύριοι, το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη για τις ψηφοφορίες αφορά την έκθεση Buchner και τον έλεγχο των εξαγωγών της μεταφοράς, της μεσητείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης. Ε, ε, Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορίου. Ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας.